Άρχεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε το απόγευμα. Μια καινούργια εμπειρία να βρισκόμαστε και πάλι σε αυτή την αίθουσα. Εκ μέρους της Προεδρίας, της DigiCom, της DigiInte, της DigiInlo. Σας καλωσορίζουμε. να περάσουμε απευθεία στη συζήτηση. Είναι δοκιμαστική αυτή η συνεδρίαση. Θέλουμε να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα, τα μικρόφωνα, ο φωτισμός, η διερμηνία. Δεν έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα τη διερμηνία σήμερα. Κανονική συνεδρίαση δηλαδή. <laughs> Θέλουμε απλώς, <laughs> είμαστε πάντα ευγνώμονε για την ποιότητα της, των υπηρεσιών που προσφέρεται. Αλλά απλώ κάνουμε μια δοκιμή σήμερα. Εντάξει. Θα έχετε δει όλοι το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε με μερικέ συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα για την ε, συντήρηση του Λαβρακίου και τον, το σκουμπρί του Βόρειου Ατλαντικού. Διαλέξαμε αυτές τις ζητήσεις για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί τα θέματα είναι συναρπαστικά που θα σα κρατήσουν σε γρήγορση όλα τα απόγευμα. Αλλά μην ασχοληθείτε με το περιεχόμενο της συζήτησης, ασχοληθείτε με τα τεχνικά. to use their blue cards. We want to test the blue card function as well